Αν λοιπόν ε, συμφωνείτε μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως ε, με κάποια μικρή κατηστέρηση. μπορούμε να επαναλάβουμε τις εργασίες μας. Ε, σήμερα το πρωί είχαμε ένα πολύ έντονο πρωινό. Είχαμε εδώ τέσσερις υπουργούς, Έλληνες υπουργούς, οι οποίοι μας ε, παρουσίασαν ένα έντονο πρόγραμμα και πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους ε, επόμενους μήνες. Ξαναξεκινάμε λοιπόν τις εργασίες της Επιτροπής μας με την ε, εξέταση τροπολογιών ενός πολύ ενδιαφέροντος θέματος που όπως ξέρετε θα ψηφίσουμε στις 24 Φεβρουαρίου στην έκτακτη Ολομέλεια του Στρασβούργου έτσι ώστε να έχουμε το χρόνο να ε, προετοιμαστούμε κιόλας ε, για τις ε, εκλογές αλλά να κάνουμε καλά και τη δουλειά μας. Έχουμε λοιπόν τη συζήτηση για τις τροπολογίες. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Πιλάρ Ντεκαστίγιο για να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες. Και κατόπιν έχουν αντικατασταθεί κάποιοι συνάδελφοι που είναι ισκιώτης Όλοι βέβαια είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι ε, και είμαι σίγουρη ότι η συζήτησή μας θα είναι υποφελής για όλους. Πιλάρ, ε, σου δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που έφτασα με κάποια καθυστέρηση, αλλά ήμουνα σε μια συνάντηση επίγουσα. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς, μπορούμε τώρα αρκετά ήρεμα να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες θα είμαι σύντομη, ξέρετε, γιατί πάνω απ' όλα θέλω να ακούσω τους συναδέρφους. Εξάλλου είχα την ευκαιρία σε διαφορετικά πλαίσια συναντήσεων με σκιώδης και στου διαδρόμου κτλ. μου δόθηκε ευκαιρία να ακούσω τις απόψεις και των συναδέρφων και έτσι να διαμορφώσω την άποψή μου για το πακέτο αυτό. Το πακέτο αυτό για την εσωτερική αγορά τηλεπικοινωνιών πρέπει να σας πω ότι κατά πρώτον πέρα από τις τεράστιες δυσκολίες χρονοδιαγράμματος βάσει των όσων παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλα αυτά αναγνωρίζω το ενδιαφέρον και την αποφασιστικότητα της Επιτροπής και ιδιαίτερα της Επιτρόπου Κρούς που δεν θέλει να αφήσει αυτή την κοινοβουλευτική θητεία να περάσει χωρίς να παρουσιάσει σύνολο μέτρων για να δώσει νέα όθηση στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τηλεπικοινωνίες, για παράδειγμα, που αποτελούν και τον βασικό πυλώνα κατά κάποιο τρόπο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και της ψηφιακής οικονομίας. Για να έχουμε μια ανάπτυξη λοιπόν της ψηφιακής αγοράς, οι ψηφιακές τηλεπικοινωνίες είναι θεμελιώδης. Από εκεί και πέρα λοιπόν θέλω να πω το εξής. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρισκόμαστε σε μια μοναδική κατάσταση και τελική φάση που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε να τελειώσει αυτή η θητεία χωρίς να συνεισφέρουμε κι εμείς στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των συνθήκων σε ένα τομέα που στο κάτω-κάτω είναι τομέας συνολικά της τεχνολογίας πληροφοριών και πιο συγκεκριμένα των τηλεπικοινωνιών. Γιατί είναι κάτι πολύ βασικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οπότε, όσο καλώς και αν ακούγεται αυτός ο στόχος στα λόγια, πέραν αυτού πρέπει να έχουμε αποτελέσματα βάσει πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι επιπτώσεις είναι μεγάλες στην αντιγωνιστικότητα των οικονομιών μας. Έχει μεγάλες επιπτώσεις επίσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Θετικές επιπτώσεις βέβαια. Γι' αυτό και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με ανοιχτό πνεύμα και με μεγάλη φιλοδοξία και επιθυμία να πετύχουμε το στόχο μας. Επί του περιεχομένου τώρα, όπως έχω πει και άλλες φορές, η πρόταση αυτή δεν πρόκειται να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς. Όχι. Θα μείνουν πράγματα να γίνουν πολλά για να έχουμε μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να γίνονται όλα online. Όμως θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντική πρόοδο και αποτελείται από επιμέρους μέτρα που όλα εφόσον τεθούν σε εφαρμογή θα έχουν θετικές επιπτώσεις, αν πάρουμε βέβαια τις σωστές αποφάσεις. Έτσι, αν δεν τις πάρουμε, όχι βέβαια. Τα μέτρα αυτά αποτελούν πυλώνες που πάνε από το ραδιοφάσμα, από τον καλύτερο συντονισμό, την βέλτιστη χρήση του ραδιοφάσματος που είναι αποφασιστική σημασίας για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και για την ανάπτυξη των ε, επικοινωνιών και της ευρυζωνικότητας. Επίσης, έχει σχέση με την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον κλάδο αυτός ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, Πρέπει να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία και να καταλήξουμε σε μια ενία αδειοδότηση για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε το γεγονός ότι ο Μπέρεκ, ο φορέας δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Ρυθμιστικών Αρχών, αποτελεί και τον φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ρύθμιση και ό,τι έχει να κάνει με τη ρύθμιση και γύρω από τη ρύθμιση δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς, ο Μπέρεκ λειτουργεί εδώ και λίγο. Ο ρόλος του πάντως είναι σημαντικός και η αναγνώριση του φορέα του Ευρωπαϊκού Ρύθμισης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και έχει να κάνει με την ίδια τη φύση του διαδικτύου. Και αυτό δεν είναι σημαντικό όπως και τα άλλα βέβαια. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε εδώ για το ότι έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το δίκτυο, το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αφήνει κανέναν απ' έξω. Αντίθετα, ενισχύει τη συμμετοχή όλων. Πάντα δίνει την ευκαιρία για συμμετοχή σε όλους. Και γι' αυτό και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας ώστε να αναπτύξουμε νέους τρόπους εκπαίδευσης, κατάρτασης, παροχής υπηρεσιών από πλευράς των κυβερνήσεων και οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία θέλει να αναπτύξει ένα μοντέλο εμπορικών συναλλαγών, για οποιονδήποτε έχει ταλέντο, δημιουργικότητα, όρεξη. Το διαδίκτυο βοηθάει οποιαδήποτε πόρτα, οποιαδήποτε στοιχείο. που περιορίζει το διαδίκτυο, έτσι κι δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, αλλά σίγουρα θα ήταν αντίθετο με την ίδια τη φύση του διαδικτύου. Γιατί το διαδίκτυο, είπαμε, είναι για όλους. Είναι για τους χρήστες, είναι για τις επιχειρήσεις, είναι για τους πολιτές, για τους αγοραστές. Το διαδίκτυο είναι για οποιοδήποτε έχει όρεξη, διάθεση, ταλέντο να μπει σε αυτό το τεράστιο δρόμο, σε αυτή τη λοφόρο, θα έλεγα πιο σωστά, που είναι η τεχνολογία του διαδικτύου. Και από εκεί και πέρα θα είναι πιο εύκολο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας, γιατί αν ε, δεχτούμε σαν δεδομένο ότι το διαδίκτυο μας συμπεριλαμβάνει όλους, είναι για τη συμμετοχή όλων και δεν αποκλεί κανέναν, θα είναι πιο εύκολο να προχωρήσουμε. Τέλος υπάρχει και περιαγωγή. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι έφτασε η ώρα, έφτασε η στιγμή να πάψει πια αυτό το κόστος με το οποίο επιφορτιζόμαστε κάθε φορά που μιλάμε με περιαγωγή στο τηλέφωνο. Είναι σημαντικό αυτό και για τους φορείς Καμιά φορά δεν υπάρχει συμφωνία με τον πάροχο τον τοπικό και το κόστος είναι ε, μεγάλο. Αν πάντως μπορεί κανείς να μην επιφορτίζεται με περιαγωγή, θα μπορεί να χρησιμοποιεί και περισσότερο για ανταλλαγή δεδομένων την περιαγωγή. Σε κάποια πράγματα πρέπει ακόμα να τα βρούμε βέβαια. Αλλά νομίζω ότι ως επιτοπλίστων συμφωνούμε. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχοντας δει τις τροπολογίες, οι οποίες είναι πολλές, αλλά εντάξει, όχι και φοβερά πολλές, πιστεύω ειλικρινά ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για συμφωνία σε όλους τους τομείς. Μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία λοιπόν. Ειλικρινά το πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε βρία στήριξη από την Επιτροπή μας αυτή και έτσι θα καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. 24 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε εδώ και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια και εκεί πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μεγάλη στήριξη. Έτσι θα φτάσουμε στον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο από το Σεπτέμβριο πια κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα καλές. Εφόσον βέβαια είμαστε ενωμένοι και η θέση μας είναι μια θέση συνοχής. Οι ευκαιρίες υπάρχουν. Όλα εξαρτώνται από εμά. Πραγματικά και κανένας δεν θα καταλάβαινε αν απορρίπταμε τις τεράστιες ευκαιρίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε η Επιτροπή μας να καταλήξει με μεγάλη στήριξη στη θέση της. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να καταλήξουμε σε μια πρόταση που να στηρίζουμε όλοι, έχοντας στο μυαλό μας ένα διαδίκτυο ανοιχτό που προτρέπει για συμμετοχή όλους και όχι ένα διαδίκτυο που αποκλείει. Οπότε είμαι πεπισμένη ότι όλοι θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο της συμμετοχής όλων στο διαδίκτυο και των ευκαιριών για όλους είναι μια τεράστια ευκαιρία για μας. Αν δεν τη χρησιμοποιήσουμε, τότε θα είμαστε υπόλογοι στους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι δεν θα καταλάβουν γιατί το κάναμε. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα θέλω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πιλάρ για αυτή την ε, ενημερωτικότατη παρουσίαση. Δεν είναι παρόντες ε, όλοι οι σκιώδεις Έχουμε τους αντικαταστάτες τους. Ε, η έντιθε είναι η αναπληρώτρια του σκιώδου ηγητού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το ότι δεν μπορεί να είναι σήμερα παρούσα η Κάθριν, αλλά μου έχει δώσει ένα κείμενο το οποίο θα ήθελα να το διαβάσω για τα βασικά θέματα να επενθυμίσω, ε, μάλλον θέλω να τα πω αυτά για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Η ενιαία εξουσιοδότηση. Αυτό κατά την άποψή μας είναι ο πιο απλός ε, συμβασμός στο η μορφή που το έχει προτείνει ο εισηγητής. Ε, επίσης περαιτέρω διευκρινήσεις και το προτείνει ο εισηγητής και συμφωνούμε και εμείς Κατά τα άλλα, όσον αφορά την ε, έκθεση, την πρόσφατη που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, εκεί προβλέπονται διάφοροι τρόποι για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία του Μπέρεκ. Ε, για το TSM υπάρχουν ε, τροπολογίες, να υπάρξει αναδιάταξη, να μετατραπεί σε έναν ε, κανονικά λειτουργούντα οργανισμό. Όμως αυτά δεν είναι αυτή τη στιγμή απόλυτα σωστά. Όλοι συμφωνούν ότι ο Μπέρεκ είναι όλο και πιο αποτελεσματικός και αυτό είχαμε σκεφτεί κατά νου όταν πρώτο ιδρύθηκε. Άρα δηλαδή θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε ριζικά τη δομή του. Και επιτρέψτε μου εδώ και μία προσωπική παρατήρηση. Από ό,τι βλέπω θα υπάρξει διάλογος ε, με τους νέους υποψήφιους για τον Μπέρεκ. Ο ένας από αυτούς είναι από τη δική μου τη χώρα και μπορώ με χαρά να σας πω ότι στο ε, Συμβούλιο έχει κάποια εμπειρία, γνωρίζει το θέμα, άρα δηλαδή υπάρχουν κάποιες εγγύησεις για την Επιτροπή ΙΤΕΡ. Το βασικό μήνυμα για τον Μπέρεκ είναι ότι δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τίποτα πριν ε, προχωρήσει ο οργανισμός αυτός. Μπορούν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά μέσα στην δομή που υπάρχει σήμερα. Όσον αφορά την, ε, τις εναρμονισμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες, ξέρουμε ότι στην Ευρώπη έχουμε ψηλές ενεργειακές τιμές που παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητά μας. Ε, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση των τελών επικοινωνίας αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, συνεργασία σε αυτό τον ε, τομέα. Και αυτό είναι η σύσταση παριθμών 9 της περσινής μελέτης ε, σχετικά με την ψηφιακή κοινωνία και εκεί ε, προτείνεται να υπάρχει κάποια ανάλυση αγοράς που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Το επόμενο που θέλω να πω, τέρκο και ούτητη, να υπάρχει ίση μεταφορά με, με, με 71, 72 72-73 νομίζω είναι τροπολογίες ε, που πρέπει να εξεταστούν ε, και αυτό είτε για να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίε EBB ή να ε, προτείνουμε την εξαίρεσή τους. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου τις αλλαγές επί των οποίων έχουμε αποφασίσει. Αυτές μπορεί να έχουν ποιοτικέ επιπτώσεις σε όλα τα άλλα νομοθετικά κείμενα, ας πούμε στην οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι λοιπόν σαφές ότι θα πρέπει να επαναξετάσουμε την ε, αλληλένδεση μεταξύ ε, της ε, την παροχή υπηρεσιών γενικότερα και την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη διευκρίνηση. Όσον αφορά το φάσμα, ε, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οφείλουμε να ενταχθούμε ε, μέσα στην τραυσοδογία και το SPP. Ισορροπία ανάμεσα στους ε, παρόχους και τους τέρκο όπως επίσης και να είναι ανοιχτή η πόρτα για την ανάλυση του φάσματος. Υπάρχουν όμως εδώ δύο νέα στοιχεία που πρέπει να έχουμε κατά νου πρώτον, ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα από την ελάχιστη διάρκεια της άδεια, περίπου 30 χρόνια, και να προσπαθήσουμε ε, ε, καλύτερη παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα και αν η Επιτροπή πρέπει να αποδείξει ότι ε, πρέπει, έχει τι αρμοδιότητες για τη διαχείριση του φάσματος. Το θέμα των παρεμβολών ε, δεν απαντάται στο κείμενο της Επιτροπής. Η Κάτριν έχει καταθέσει τροπολογίες επί του θέματος για να διασφαλίσει ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεπάρχουν χωρίς πρόβλημα. Συμφωνούμε λοιπόν με τα περισσότερα σημεία του εισηγητή. Παρόλα αυτά υπάρχουν άλλα δύο θέματα που είναι λίγο πιο προβληματικά και είναι τα δύο εξή. Πρώτον, όσον αφορά την περιαγωγή, η θέση του Κοινοβουλίου που είναι υπέρ του να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής ε, ε, δεν έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή σίγουρα ε, πολλοί θα πούν ότι το 15, το 16 πρέπει να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής. Και αν δούμε τις τροπολογίες θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν βοηθητικά μέτρα, άρα δηλαδή ποιος είναι ο σωστός τρόπος ε, να ε, προχωρήσουμε. Και με ποια ακριβώς διατύπωση πρέπει να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε για την τελική λύση. Όσον αφορά την ουδετερότητα, ε, θα πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε να εξετάσουμε τις υπηρεσίες διαδικτύου ε, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και επίση ε, και τις ε, προδιαγραφές για το τι είναι λογική διαχείριση. Στις εξειδικευμένες υπηρεσίες να υπάρχει αναφορά σε κλειστά δίκτυα. Αυτό αναφέρεται σε ε, πολλές ε, τροπολογίες και δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Σε επίπεδο της διαχείρισης της κυκλοφορίας, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει κλειστός ή ανοιχτός κατάλογος κριτηρίων, τώρα εξετάζουμε το σχέδιο ε, των τροπολογιών συμβιβασμού. Είναι πολύ μεγάλο το έργο αυτό, γι' αυτό Πιλάρ σου ευχόμαστε καλή τύχη και εμείς είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Το λόγο συνάδελφος Ρόντε από τους φιλελεύθερους. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα σήμερα. Δεν θέλω να πω πολλά. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι δεν βρήκα τίποτα μέσα στην έκθεση της Πλέρ με το οποίο να μην συμφωνώ. Όντως, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν κάτι το οποίο θα προσφέρει μια πραγματική προστιθέμενη αξία στους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνουμε εμείς αυτή τη διαφορά. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτή την τελευταία εκδοχή που μας παρουσίασε σήμερα η Πιλάρα. εδώ και 9 μήνες, έτσι κι συμφωνούσαμε με τις κύριες κατευθύνσεις. Από εκεί και πέρα δούλεψε πάρα πολύ η Πιλάρ. Και αυτό που μας παρουσίασε σήμερα συμπεριλαμβάνει τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες συμφωνήσαμε. Υπάρχουν επίσης δύο τομείς όπου η ομάδα μου υπέβαλε τροπολογίες. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της ημερομηνίας για την περιαγωγή. ...2015 πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι. Και γιατί τώρα, όχι γιατί κάποιοι λένε 2016, αλλά γιατί αν όλα αυτά τα θέματα τιμής συνεχίσουν να συζητιόνται μέχρι το 2016, τελικά η πρόταση θα πρέπει πριν να μας έχει κάνει την πρότασή της η Κομισιόν, αλλά δεν θα προλάβουμε να θέσουμε τίποτα σε εφαρμογή για την κατάργηση του roaming μέχρι το 2016. Εφόσον υπάρξει η απαγόρευση αυτή της παιδιαγωγής, ή εν πάση περιπτώσει η εν περιπτωσει η απαγορευση της πληρωμής για την περιαγωγή και όταν θα έχουμε τις λεπτομερείς προτάσεις, τότε και εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε με τη χονδρική πώληση. Και εκεί θα πρέπει να βάλουμε κάποια οροφή, γιατί αν δεν βάλουμε οροφή για τη χοντρική πώληση, τότε θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε πέντε μεγάλα μονοπόλια, πέντε δηλαδή πρωταγωνιστές, τηλεφώνικα, την ε, Orange κλπ. Αυτοί θα μείνουν στο παιχνίδι, γιατί αυτοί διαθέτουν ήδη τις υποδομές. Αν λοιπόν σε αυτό το θέμα της χοντρικής πώληση θέλουμε οι μικροί να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους μεγάλους, τότε οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν και αυτές να στέλνουν το λογαριασμό στους πολίτες τους. Αλλιώς θα υπάρξει στρέβλωση στην αγορά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια αγορά όπου να υπάρχουν και οι μικροί και οι μεγάλοι για να υπάρχει ο καλύτερος δυνατόν ανταγωνισμός. Αυτή λοιπόν η κατάργηση της ε, περιαγωγής, της πληρωμής για την περιαγωγή, πρέπει να έχει και κάποια όροφη όσον αφορά τις χοντρικές τιμές. Και πρέπει να προβλέψουμε ως ημερομηνία την 1η Ιουλίου του 2015. Εμείς αυτή την ημερομηνία θέλουμε. Τότε θέλουμε να σταματήσει η πληρωμή για την περιαγωγή. Από εκεί και πέρα οι πολίτες δεν θα πρέπει να πληρώνουν ό,τι πληρώνουν σήμερα όταν χρησιμοποιούν με περιαγωγή τα κινητά τους. Έρχομαι τώρα στο ραδιοφάσμα. φαίνονται πιο φιλόδοξα εδώ αυτά που ζητάει η Πιλάρ από ό,τι μας έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ λοιπόν έχω υποβάλει τροπολογίες που πάνε ακόμα πιο μακριά τουλάχιστον. Εγώ το λέω αυτό. Το πιστεύει και ο συνάδελφος Ρόκμαντ μάλιστα. Και ελπίζουμε όλα αυτά να καταλήξουν. Κανείς δεν θέλει να υπάρχει διαφοροποίηση πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα ραδιοφάσματα 700-800 MHz και να δούμε και το, που, την πολιτιστική διάσταση. Όμως δεν υπάρχει εδώ αντίφαση, παρόλο που μερικοί θέλουν να βλέπουν αντίφαση εδώ. Ακόμα και αν υπάρχει ψηφιοποίηση και δεν χρησιμοποιούμε ολόκληρο το φάσμα για ε, τις εκπομπές, δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί το πολιτιστικό περιεχόμενο. Όχι, αυτό έχει ήδη βρει τη θέση του. Και στη σημερινή εποχή. Άρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι και να έχουμε αρκετό θάρρος να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες στο κάτω-κάτω θα είναι υπέρ του καταναλωτή. και θα του δείξουμε έτσι ότι του προσφέρουμε μια προστιθέμενη αξία. Επίσης πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι γιατί έτσι έχουμε μια φιλόδοξη ψηφιακή Ευρώπη, κάτι το οποίο είναι πολύ καλό για την ανταγωνιστικότητά της στον κόσμο. Και θα δημιουργηθούν και θέσεις απασχόλησης επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σκιώδης για την ομάδα της τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πιλάρτα Καστήλιο για την εκτενέστατη και περιεκτικότατη παρουσίαση του πακέτου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο σκιώδεις εισηγητές των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελεύθερων για τα σχόλιά τους και όλους για τις τροπολογίες. Τα δικά μου σχόλια δεν θα είναι ε, τόσο εκτενή. Θα αναφερθώ κυριότερα στις ε, γενικότερες διατάξεις. Πιστεύω πως ε, ήδη πάρα πολλά σημεία έχουν καλυφθεί από την πρόταση και ήταν πάρα πολύ χρήσιμος ο καταμερισμός των εργασιών όσον αφορά την εξέταση τροπολογίων. Τώρα, όσον αφορά τις συγκεκριμένες ε, τροπολογίες, ε, η τροποποίηση ενός ε, θέματος είναι πάντα κάτι το περίπλοκο. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε ορισμένες πάρα πολύ χρήσιμες τροπολογίες. Θα ήθελα να αρχίσω με ορισμένες, ορισμένα σχόλια για την βελτίωση των υποδομών των τηλεπικοινωνιών και με τις σχετικές τροπολογίες. Καταρχάς, θεωρώ πολύ χρήσιμο τον διαχωρισμό των ε, λειτουργιών. Αυτό είναι κάτι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ ε, συχνά παλαιότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω πως αυτός ο λειτουργικός διαχωρισμός θα είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και έτσι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να εστιάσουν με, ε, στο να δώσουν κίνητρα για καλύτερες επενδύσεις σε περισσότερη ευρυζωνική τεχνολογία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, με χαρά μου βλέπω ότι συνεχίζουμε να έχουμε προτεραιότητα για την ε, αποδέσμευση. Βλέπω ότι στηρίζεται αυτό από πολλές ε, πολιτικές, ομάδες και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν οι πολίτες πρόσβαση στις βριζονικές ε, υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ το ΕΛΚ για την πρόταση της κατάργησης των τελών Ιδιαίτερα ε, μία τροπολογία του κυρίου Βανίστελροι αναφέρει ότι χρειάζεται, ε, χρειάζονται καλές επενδύσεις και πρόσθετα μέτρα στον τομέα αυτό. Και αυτό επίσης θεωρώ πως θα είναι ε, καλό και για όλον τον κλάδο και όπως ανέφερε και ο κύριος Ρόντα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος για το μέλλον της ευρυζωνικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, με χαρά μου βλέπω ότι υπάρχει ευρεία στήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες για το ανοιχτό διαδίκτυο. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον ορισμό του. Πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχει από πίσω ένα κλειστό δίκτυο επιπλέον. Το ανοιχτό δίκτυο είναι κάτι που ευνοεί πάρα πολύ την ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα στον τομέα των τεχνολογιών και αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ ισχυρή, ιδιαίτερα στα πλαίσια της ψηφιακής αγοράς. Έπειτα, ε, το τι ακριβώς είναι ένα κλειστό δίκτυο είναι κάτι που θα επεξεργαστούμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των ε, σχεδόν εισηγητών. Πέραν αυτού όμως πιστεύω πως έχουμε εδώ μια πάρα πολύ καλή βάση για να ε, επιτευχθεί μια συμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες, διότι όλοι επιθυμούμε μια καινοτόμο πλατφόρμα όπου όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες. Ε, με αφορμή αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στις εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται από αρκετές πολιτικές ομάδες και τις ε, οποίες συζητούν και άλλες επιτροπές. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα των εξειδικευμένων υπηρεσιών φαίνεται να είναι η δυσκολία στο να ορίσουμε τι ακριβώς είναι αυτές οι εξειδικευμένες υπηρεσίες και ποιος θα τις παρέχει. Έχω δει πολλές τροπολογίες οι οποίες ε, κατευθύνονται στις υπηρεσίες ε, της κοινωνία των πληροφοριών, στην καινοτομία και στη σύνδεση των ε, υπηρεσιών που χρησιμοποιούν την υποδομή των τηλεπικοινωνιών για να ε, συνδέσουν τους ε, πολίτες. Επίσης, όντως δεν, υπάρχουν, δεν είναι σωστά ρυθμισμένος ο τομέας αυτός και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό, χρειάζεται περισσότερη ρύθμιση, ωστόσο χρειάζεται επίσης και προσοχή οι υπηρεσίες αυτές να ρυθμίζονται στα πλαίσια των ε, τηλεπικοινωνιών, των κανονισμών και της τηλεπικοινωνίες. Χρειαζόμαστε επομένως μία ε, περιεκτικότερη έρευνα και έκθεση για το ποιοι τομείς είναι εκείνοι που θα υποφεληθούν περισσότερο από περισσότερο έλεγχο και επίσης να εστιάσουμε στα συγκεκριμένα ε, σημεία, διότι δεν μπορούμε να είμαστε γενικοί και να καλύψουμε με ένα άρθρο τα πάντα. Ε, η κυρία Χέρτσοκ ζήτησε μια ανεξάρτητη εκτίμηση αντικτύπου που θα οδηγήσει σε μια ανεξάρτητη επίσης πρόταση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ε, υπηρεσίες αυτές και πιστεύω πως στην Επιτροπή θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και σε αυτό. Επίσης, ε, είναι σημαντικό να αποφύγουμε την υπερβολική γραφειοκρατία, διότι αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη ασάφεια για όλους τους ενδιαφερόμενους της αγοράς, Ιδιαίτερα στον ε, τομέα Voice IP υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ασάφεια και πιστεύω πως αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή ε, και από τους συνομοθέτες και από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τέλος, θα, θα ήθελα να στηρίξω ορισμένες από τις ε, τροποποίησεις και τις προτάσεις των φιλελεύθερων. Πιστεύω πως ε, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα. Και επίσης να δώσω την πλήρη στήριξή μου για την ε, πρόταση περί φάσματος χωρίς άδειες που υπέβαλαν οι σοσιαλδημοκράτες. Να πω επίσης ότι αυτό ότι αυτός ο τομέας είναι ο τομέας όπου έχουμε τις ε, ε, μεγαλύτερες καινοτομίες. Αντίθετα με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης των τεχνολογιών φάσματος. Και πιστεύω πως εδώ έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες για καλές και σύγχρονες ε, επενδύσεις, τις οι οποίες θα μας ε, βοηθήσουν και θα τονώσουν την ε, αγορά μας. Θα, μπορούσαμε επίσης να, θα μπορούσαν επίσης να χορηγηθούν ορισμένες άδειες για συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένες τεχνολογίες του φάσματος. Αυτά από μένα θα χαρώ να συνεργαστώ με τους υπόλοιπους κοιόδης εισηγητές. Κύριε και αυτός και ο εισηγητής έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρωτού συζητήσω τις τροπολογίες ε, λεπτομερέστερα θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένος με τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αρμόδιου Επιτρόπου. Δεν απάντησαν ούτε στην προφορική ερώτηση η οποία ετέθη στην ε, Ολομέλεια, ούτε στη γραπτή ερώτηση, την οποία έστειλα έπειτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το βρίσκω αυτό αρκετά περίεργο το να μην λάβω καμία απολύτω απάντηση. Τώρα, όσον αφορά τι τροπολογίε, να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια για όλη την δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα και την ε, επιτυχημένη συνεργασία και να της δώσω επίσης και τη στήριξή μου και για την έκθεση και για τις τροπολογίες. Ωστόσο, αισθάνομαι ότι χρειάζεται περισσότερη εξέταση, περισσότερη αναθεώρηση του ε, για το φάσμα. Έχουμε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συγκεντρώσει ε, την ε, εξουσία, τη ρυθμιστική εξουσία και να μην δώσει την εξουσία αυτή στα κράτη-μέλη. αναθεώρηση λοιπόν και συντόμευση του κειμένου. Τώρα, ως, επίσης, ε, θεωρούμε πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί, να διευκρινιστούν οι ορισμοί στην πρόταση. Εμείς προτιμούμε την διατύπωση του συναδέλφου κυρίου Χάρμπορ στην γνωμοδότησή του από την Επιτροπή, της Επιτροπής Υπάρχουν μικρές διαφορές. Και τώρα όσον αφορά τον στόχο της περιαγωγής. Κανεί δεν θα ήθελε να καταργηθεί η αγωγή περισσότερο από εμένα. Και το συντομότερο δυνατόν μάλιστα. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε τι πραγματικά μπορεί να γίνει. Δεδομένου ότι μόλις τώρα έχουμε τελειώσει ε, το νομοθετικό μας έργο για την περιαγωγή, το να προχωρήσουμε παραπάνω είναι κάτι που χρειάζεται πρώτα μία περίοδο προσαρμογής. Η κυρία Ντεκαστήγιο πρόσφατα μας ε, ανέπτυξε τους ε, λόγους για τους οποίους ε, θεωρεί το 2005 στόχο, χρονικό σημείο για το, στο οποίο θα καταργηθεί η περιεγωγή. Πολύ ωραία θα ήταν στη θεωρία, αλλά στην πράξη το θεωρώ μη εφικτό. Και νομίζω πως το 2016 θα ήταν κάτι πιο ρεαλιστικό. Ευχαριστώ. Τελείωσαν λοιπόν οι παρεμβάσεις των ε, σχεδόν και έτσι θα ξεκινήσουμε με τις ε, παρεμβάσεις των ε, συναδέλφων που είναι δυνατόν παρακαλώ να περιστούν σε τρία λεπτά. Ο συνάδελφος Χόκμαρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους τους άλλους που παρενέβησαν. Αν δούμε λιγάκι τις ε, τροπολογίες θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ε, αρκετές ε, τροπολογίες και νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ε, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια βήματα προς τα εμπρός. Κάτι που άκουσα τους τελευταίους μήνες είναι το εξής. Μερικές φορές η συζήτηση γίνεται για το κατά πόσον η Ευρώπη καθυστερεί και κατόπιν γίνονται συζητήσεις που κατατείνουν στο ότι δεν ε, υπολοιπόμεθα. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά δεν έχουν νόημα γιατί αν δει κανεί το γεγονός ότι η Ευρώπη στο σύνολό της οικονομία υπολείπεται δεν νομίζω ότι ε, αμφισβητεί κανείς ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Και αυτό λόγω του ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, οι τηλεπικοινωνίες και η ψηφιακή επικοινωνία για την ε, ανταγωνιστικότητα, κυρίως στο μέλλον. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι είμαστε τόσο καλοί όσο και, όλο, οι άλλοι στον τομέα αυτό, τη στιγμή που ε, καλούμεθα να είμαστε συνεχώς καλύτεροι. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθούμε ταχύτερα κατά τα επόμενα χρόνια. Αν δούμε λιγάκι τις ε, τροπολογίες και τις ε, προτάσεις ε, του εισηγητή που σε τις μάλλον σε μεγάλο βαθμό στηρίζω και στις λεπτομέρειές τους, το θέμα είναι να είμαστε ρεαλιστικοί και παράλληλα αποφασιστικοί. Με την έννοια ότι θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και θα επιφέρουμε περισσότερες καινοτομίες σε αυτή την αγορά. Θα κάνουμε βήματα προς τα εμπρός, προς την κατεύθυνση της ε, ενέας ε, αγοράς. Αυτό λοιπόν πρέπει να ορίσουμε ως στόχο. Ο συνάδελφός μας, ο κύριος Τσίτσεστερ, τον οποίο τον στηρίζω γενικά, αλλά και σε πιο ειδικά θέματα, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα παράδοξο όσον αφορά την περιαγωγή και το να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι εφόσον επιμένουμε ότι αυτή η αγορά πάνω από όλες πρέπει να παραμείνει εθνική, τότε ενδέχεται να προσφερθεί η δυνατότητα να προχωρήσει κανείς με διατίμηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ε, αποτινάξει την περιεγωγή. Μόνο τα τέλη περιεγωγής μπορεί να αποφύγει. Γιατί όσο υπάρχουν 28 διαφορετικές αγορές ε, θα παραμένει περιεγωγή με όλες τις συνέπειες. Αυτό λοιπόν πρέπει κανείς να το έχει κατά νου. Και θέλω να πω ότι όσον αφορά το φάσμα Πρέπει να προχωρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη το τι αποφασίστηκε στο πρόγραμμα ραδιοφάσματος. Να οριστούν οι στόχοι, αλλά επίσης να ανοίξει το ραδιοφάσμα λόγω του ότι είναι στρατηγική σημασίας να υπάρχουν οι δυνατότητες μεγάλης ταχύτητας που είναι καθοριστική σημασίας για το μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι είναι αναπόφευκτο να συζητήσουμε και την απαγόρευση 700 ban, αυτό που πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον. Το δεύτερο αφορά το φάσμα πάλι. Νομίζω ότι η ρεαλιστική προσέγγιση είναι να μην χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως εναρμόνιση παραδείγματος χάρη, αλλά συντονισμό και αδεία, εξουσιοδότηση, αδειοδότηση μάλλον, ε, για να μπορούμε να καταλήξουμε ενδεχομένω σε πανευρωπαϊκές λύσεις. Και αυτή είναι η τρίτη μου παρατήρηση. Όσον αφορά την περιεγωγή αυτή καθεαυτή, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα για το κατά πόσο είναι απαραίτητο ή όχι να αποφύγουμε το υψηλό κόστος της περιαγωγής. Και υπάρχει το εξής ε, περίεργο. Αυξάνονται, αυξάνεται κατά πολύ ο όγκος των δεδομένων. Η τιμή και το κόστος για τον πολίτη θα αυξάνεται όσο και αν ρυθμίζουμε το θέμα των τιμών. Γιατί η ταχύτητα και ο όγκος ε, αυξάνονται πολύ περισσότερο από τον ρυθμό με τον οποίο εμείς ε, ρυθμίζουμε τις τιμές. Και εγώ δεν πιστεύω ότι η ρύθμιση των τιμών και βραχυπρόσμα αλλά και μέσω πρόθεσμα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Το πιο σημαντικό είναι ε, να ρυθμίσει κανείς αγορές, ε, να εξαναγκάσει τους ε, παρόχους ε, να επιτρέψουν τον ανταγωνισμό. Και αυτό είναι καθοριστική σημασία και για το επίπεδο ανταγωνισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω είναι εντυπωσιακό και αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι αν δει σήμερα τις ευρωπαϊκές αγορές θα διαπιστώσει ότι οι προκλήσεις ε, κατά κύριο λόγο ε, μειώνουν τις τιμές, όχι οι κύριοι πάροχοι, αυτοί παραμένουν στο επίπεδο ε, των τιμών που έχουν ρυθμιστεί. Οι προκλήσεις είναι εκείνες που αναγκάζουν ε, στο να υπάρξει πρόοδος. Άρα δηλαδή πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ε, ανταγωνιστές, οι πάροχοι μάλλον ανταγωνίζονται μεταξύ τους τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, όσον αφορά τώρα την ουδετερότητα των δικτύων, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο θα εξελιχθεί κατά τα επόμενα έτη ταχύτατα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην ρύθμιση του διαδικτύου. Άλλο το να ρυθμίσει κανείς την πρόσβαση, την δυνατότητα να έχει κανείς ε, ε, μικρότερες ποσότητες και άλλο το να ρυθμίζει κανείς τον όγκο. Ε, και να πω τελειώνοντας, ε, σε αυτό τον τομέα χρειαζόμαστε συντονισμό, αδειοδοτήσεις ε, και να δούμε και πώς θα ενισχύσουμε τον φορέα Μπέρεκ. Όχι επειδή εδώ έχουμε τον υποψήφιο εκτελεστικό διευθυντή, αλλά διότι ο φορέας αυτός πράγματι θα καταστεί καθοριστική σημασία στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τις ευρωπαϊκές αγορές. Η κυρία Νίμπλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια και όλους τους υπόλοιπους ε, σχεδόν για τις ανθρωπολογίες που κατέθεσαν οι οποίες εμπλουτίζουν την έκθεση και μας δίνουν τροφή για σκέψη και για συζήτηση. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην ουδετερότητα του διαδικτύου και να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Διάβασα τις ε, σχετικές τροπολογίες για την ουδετερότητα του διαδικτύου. Υπήρξαν ορισμένες προτάσεις διατύπωσης από την Επιτροπή Πολιτισμού, ε, το πώς μπορούμε να ορίσουμε καλύτερα τις ε, υπηρεσίες και ότι φάνηκε ότι χρειαζόμαστε έναν καλύτερο και σαφέστερο ορισμό. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε φυσικά είναι να κάνουμε ένα διαδίκτυο δύο ταχυτήτων, προ, ε, πρώτης και δεύτερης θέσεις. Ε, γι' αυτό ίσως χρειάζεται και να δούμε και την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ πιστεύω πως ε, δεν πρέπει να απομακρυνθούμε πάρα πολύ και να φροντίσουμε να οδηγηθούμε σε έναν καλό συμβιβασμό. Διάβασα επίσης και τις προτάσεις των ε, συμπατριωτών μου, ιδιαίτερα από την Επιτροπή ενέργειας που ανέφεραν αυτές το διαδίκτυο δύο ταχυτήτων. Και αναφέρονται στο ότι πρέπει να αποφύγουμε να εμποδίζουμε τους ε, παρόχους τηλεπικοινωνιών και να τους ε, οδηγήσουμε σε μείωση κερδών. Ε, το σημαντικό είναι να υπάρχει παροχή στο διαδίκτυο για όλους, να μην υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δύο τάξεις ε, υπηρεσιών και να αποφευθούν έτσι αυτά τα σενάρια τρόμου που ακούμε τώρα τελευταία στο γερμανικό τύπο για το διαδίκτυο. Έπειτα, αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι κάτι που έχει να κάνει με, ε, το σύνολο της ε, πρότασης και θα σας μιλήσω ειλικρινά. Εδώ έχουμε συζητήσει πολλές ε, φορές για όλη την βιομηχανία τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, για το μέλλον της, για τις νεότερες εξελίξεις, ιδιαίτερα από την πλευρά της Ανατολικής Ασίας και ο στόχος μας φυσικά είναι να ανακάμψει η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, Κίνα και την Νότια Κορέα. Και αυτό που προέχει είναι να φροντίσουμε ο τομέας ε, ICT να ανακάμψει, να βελτιωθεί, έτσι ώστε να βελτιωθεί και η κατάσταση της ε, δικής μας ε, βιομηχανίας. Τώρα όσον αφορά την ε, περιαγωγή, πιστεύω πως οι υπόλοιποι συνάδελφοι τα είπαν όλα, έχουν απόλυτο δίκιο. Αυτό το πρόσθετο κόστος είναι επιζήμιο για τις εταιρείες μας, για τη βιομηχανία μας. Και όσον αφορά τις ε, συχνότητες και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, αυτό φυσικά είναι ένα πρόβλημα και θα επιδεινωθεί. Ιδιαίτερα με, τους, ε, με τις ε, μεγάλες εταιρείες, με την Nokia, με την Ericsson, με, αυτή την συγκεντρωτική τάση που έχει παρατηρηθεί. Ήδη είχαμε πριν από μερικά χρόνια το πρόβλημα με τις συχνότητες GSM των κινητών τηλεφώνων. Και αυτό δεν φυσικά πρέπει να συνεχιστεί. Είναι κάτι που σχετίζεται και με πάρα πολλούς ε, τομείς. Αυτές ε, ήταν οι κάπως πιο γενικές παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Φυσικά υπάρχουν λεπτομέρειες ε, τις οποίες θα συζητήσω. Σίγουρα χρειάζεται στήριξη της βιομηχανίας. Όμως σε κάθε περίπτωση πιστεύω πως αυτή εδώ η Επιτροπή είναι το καταλληλότερο φόρουμ για να γίνουν σωστές προτάσεις. Και πιστεύω πως οι περισσότερες προτάσεις που έχουν γίνει είναι οι σωστές. Δίνω το λόγο στον κύριο Ζαλέσκι ε, που ήταν και σήμερα το πρωί εδώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να μιλήσω όμως πολωνικά αν μου επιτρέπετε. Πρέπει να σας πω ότι ακούγοντας την ε, παρουσίαση της Πιλάρ ακούσαμε την φιλοσοφία. Ο κόσμος των τηλεπικοινωνιών εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Συνεπώς πρέπει να αντιδράσουμε και εμείς γρήγορα στις χώρες. Μη μέλη το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Ξέρουμε πόσο πολύ θέλουμε μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά μεγαλύτερη ελευθερία σημαίνει και μεγαλύτερο κίνδυνο για το πώς θα δράσουν οι άνθρωποι και μερικές φορές τα αποτελέσματα δεν τα περιμένουμε, είτε πρόκειται για πάτες, είτε πρόκειται για τρομοκρατία. Απάτες και στην επιστημονική έρευνα, μεταξύ άλλων. Συνεπώς πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Ο κύριος Τσίτσεστερ είπε ότι να είμαστε πιο ενωμένοι, αλλά να μην υπάρχει κεντρική διαχείριση. Χρειάζεται κάποια ρύθμιση που να βασίζεται στο συντονισμό. Αυτό μπορεί να κάνει το ευρωπαϊκό επίπεδο και αν αυτό το τραβήξουμε λίγο πιο πέρα. Όταν έχουμε θέματα εθνική ταυτότητας κλπ. Δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε. Όταν όμως μιλάμε για τις τηλεπικοινωνίες, εδώ είναι ένας τομέας που όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δράσουμε από κοινού. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θέλουμε να αγνοήσουμε τις διάφορες αξίες μας. Πρέπει να εξυπηρετούνται κοινά συμφέροντα με ό,τι κάνουμε. Τώρα υπάρχει κάποια αντιπαράθεση εδώ, γιατί έχουμε τους πάροχους υπηρεσιών που προσπαθούν να μας κάνουν να υποφελθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Ναι, αλλά θέλουμε φτηνή πρόσβαση στο διαδίκτυο συγχρόνως για κάθε πολίτη. Αν λοιπόν τεχνολογικά τα λύσουμε όλα, αν υπάρχει ασφαλής πρόσβαση, τότε πιστεύω ότι και οι επιχειρήσεις και όλοι θα υποφεληθούν. Από την πιο εύκολη δηλαδή και απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουμε από τον ακαδημαϊκό κόσμο, συνήθως κάνω διαλέξεις. Όταν επέστρεψα από την Καλιφόρνια, τη δεκαετία του 90, δεν ξέραμε καλά καλά τι να κάνουμε με το διαδίκτυο, στέλναμε mails. Τώρα βέβαια τα πράγματα πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα, η τεχνολογία επίσης εξελίσσεται πολύ γρήγορα και γι' αυτό λέω ότι πρέπει και εμείς να διασφαλίσουμε ότι έχουμε την τεχνολογία εχμής με την ασφάλεια βέβαια που απαιτείται. Γιατί τα χρησιμοποιούμε για την εκπαίδευση. Δείτε τα 14 χρόνια τι κάνουν με το διαδίκτυο. Οι νέοι φτιάχνουν ομάδες και συνομιλούν μεταξύ τους. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι για παράδειγμα δεν φορτώνουν παράνομα πράγματα, γιατί αυτό είναι αδίκημα. Άρα υπάρχει και η πτυχή της εκπαίδευσης, της διαπαιδαγώγησης σε ένα, τομέα, που η πρόοδος και ανάπτυξη είναι τεράστια και ταχύτατη. Δεν ζούμε μόνο μέσα στην Ευρώπη, ζούμε και στον ευρύτερο κόσμο. Άρα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες, αλλά και ποιες είναι οι ενδυνάμει καταχρήσεις που μπορεί να γίνουν στον κόσμο. Πιλά, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ για το εξαίρετο έργο σου. Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα πολύ καλό εγγραφό. Συνεκτικό. Γιατί σημαίνει ότι μπορεί κανείς να το διαβάσει γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πατρίσια. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, την Πιλάρτε Καστίγιο και έχω να κάνω λίγα σχόλια, επιτρέψτε μου. Έχω υποβάλει πολλές τροπολογίες, είναι αλήθεια. Και στην πραγματικότητα, στόχος του εγγράφου αυτού θα έπρεπε να είναι η εναρμόνιση και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περίμενα με πολύ ενδιαφέρον την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι από τη μια περίμενα να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής και ήλπιζα ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που να μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Ελεκτρονικών επικοινωνιών. Ήθελα λοιπόν την κατάργηση του τέλους περιαγωγής, να έχουμε τις ίδιες τιμές δηλαδή, όπως και για τις επικοινωνίες που γίνονται μέσα σε μια χώρα. Αφετέρου όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίμενα και τα διαρθρωτικά μέτρα στα οποία είχαμε αναφερθεί όταν πριν από μερικά χρόνια εγκρίναμε τον κανονισμό για την περιαγωγή. Όμως, κατά τη γνώμη μου, η πρόταση αυτή προσπαθεί να λύσει υπερβολικά πολλά πράγματα και μάλιστα με έναν τρόπο που νομίζω ότι επιδέχεται βελτίωση. Η πρόταση δηλαδή πιστεύω ότι δεν θεμελιώνεται ικανοποιητικά σε διάφορα σημεία. Για παράδειγμα, για τους Ευρωπαίους φορείς. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν είμαι κατά των Ευρωπαίων φορέων, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να τους προσφέρουμε μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση από ό,τι τους εθνικούς φορείς. Οπότε, προσπάθησα πραγματικά από την νομοθετική πρόταση να αφαιρέσω τις διατυπώσεις εκείνες που προτείνουν οι Ευρωπαίοι φορείς να μην πληρώνουν ε, φόρους, ενώ εθνικοί πληρώνουν. Αν λοιπόν εδώ θέλουμε να μιλήσουμε για την αρχή της μη διάκρισης που να διασφαλίζεται ε, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε από την άλλη ένα πλαίσιο πιο ευνοϊκό για τους ευρωπαίους φορείς. Το ίδιο ισχύει και για το ραδιοφάσμα. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, πριν από από λίγο καιρό εγκρίναμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το ραδιοφάσμα. Φροντίσαμε να θέσουμε προθεσμίες, στόχους και ήδη τότε ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο. Γιατί όλοι το ξέρουν, τα κράτη-μέλη πιστεύουν πως το ραδιοφάσμα είναι εθνική αρμοδιότητα. Είμαστε λοιπόν υπέρ της εναρμόνισης και θέλουμε να ενθαρρύνουμε την εμφάνιση νέων καινοτόμων υπηρεσιών. Όμως η πρόταση νομοθετικού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να βελτιωθεί και σε αυτό το τομέα. Και ολοκληρώνω με το εξή. Όσον αφορά το σύστημα γενικής αδειοδότησης, και πάλι κατά τη γνώμη μου, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο γενικής αδειοδότησης, αλλά πιστεύω ότι το κείμενο δεν ικανοποιεί επαρκώς και θα συμφωνήσουν φαντάζομαι και οι συνάδελφοι ότι μπορούμε να διατυπώσουμε καλές συμβιβαστικές τροπολογίες που να βελτιώνουν τις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας. Και προσθέτω μάλιστα ότι ίσως είναι μία από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τις πιο σημαντικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή την περίοδο που είμαστε στα τέλη της κοινοβουλευτικής θητείας. Οπότε, όπως και για όλες τις μεγάλες πρωτοβουλίες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και εδώ θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θα έχει να κάνει με τη ζωή κάθε πολίτη. Ακόμα δηλαδή και αν μας πάρει παραπάνω χρόνο για να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες, αξίζει τον κόπο να καταλήξουμε σε ένα απλό κείμενο που να συνεισφέρει στην ε, δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Γκέρεκ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. δεν εξέτασαμε τόση λεπτομέρεια τα θέματα αυτά, όσο εσείς όμως παρατηρώ ότι εργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και όσον αφορά τις ε, χώρες αυτές που είτε είναι γειτονικέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο θέμα της ε, ευρυζωνικότητας ιδιαίτερα στις περιοχές ε, που συνορεύουν με τρίτες χώρες, έχω να κάνω την εξή ερώτηση. Τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα, όταν βρίσκεται για παράδειγμα κάποιος στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας, τι γίνεται εκεί. Ποιον πάροχο χρησιμοποιεί κανείς τον Ουκρανικό, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. ή όταν για παράδειγμα βρίσκεσαι στα σύνορα με την Λευκορωσία, με την ε, Ρωσία. Είναι θέμα περισσότερο φυσικής. Σε ποιο δίκτυο βρίσκεσαι, σε ποιο δίκτυο χρησιμοποιείς. Τώρα και κάτι άλλο επίσης τεχνικό. Έχουμε λοιπόν ένα φάσμα το οποίο επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα στο μέλλον για μεταφορά δεδομένων, και να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις και πιστεύω ότι αυτά τα 20-30 χρόνια είναι υπερβολικά πολλά και ίσως θα έπρεπε να μειώσουμε αυτή τη χρονική περίοδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο την ε, καινοτομία στο χώρο της τεχνολογίας και η αγορά επίσης θα μπορέσει να επωφεληθεί αν χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο φάσμα το συντομότερο δυνατόν. Αυτά προς το παρόν από εμένα για το θέμα αυτό. E Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις ε, των Ευρωβουλευτών και πριν απαντήσει η συγγήτρια η κυρία Αντωνιβέλλαν από την Επιτροπή θα λάβει το λόγο για να απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις που κατ' ουσίαν αφορούν την ίδια. Ο κύριος, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήδη έχω αναφερθεί στο θέμα αυτό και στο παρελθόν. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη δουλειά της αλλά και σε όλους τους κοιόδης εισηγητές, σε όλο το επιτελείο που ασχολούνται τόσο ενεργά και συνεισφέρουν τόσο πολύ στην ολοκλήρωση της θέσης της Επιτροπής για την έκθεση αυτή. Και αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των ε, τροπολογιών. Είναι πάρα πολλές και δείχνουν αν όχι την ε, ποιότητα τουλάχιστον το ενδιαφέρον των ε, συναδέλφων για το θέμα αυτό. Τώρα θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά όσον αφορά την ενιαία εξουσιοδότηση. Σημείωσα την πρόταση της εισηγήτριας σχετικά με την εξουσιοδότηση και την απόσυρση αυτής. Μου φαίνεται πως ε, υπάρχει μια αναγνώριση του πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και φαίνεται πως αυτή η αναγνώριση εκφράζει και πολλά μέλη αυτής της Επιτροπής η θέση σας δεν είναι και τόσο διαφορετική από την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αλλά η συνεισφορά σας είναι πάρα πολύ σημαντική για να έχουμε μια εξισορροπημένη πρόταση. Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός ρόλος στη χορήγηση και ανάκληση των εξουσιοδοτήσεων θα θέλαμε να είναι ισχυρότερος. Τώρα, όσον αφορά το φάσμα, έχουμε ήδη σημειώσει την στήριξη της εισηγήτριας και πραγματικά συμφωνούμε και με τις ε, συνοδευτικές προτάσεις που αφορούν την διάρκεια του ε, φάσματος και το πόσο προβλέψιμο που είναι αυτό. Αυτό συνδέεται άμεσα με την ε, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καινοτόμων τεχνολογιών και με την ε, αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Τώρα όσον αφορά την ε, εξισορρόπηση των, ε, της ευρυζωνικότητας και των μεταδόσεων, εμείς θα θέλαμε μια καλύτερη διαδικασία συντονισμού για το φάσμα. Και να μην κρίνουμε, ε, να μην αποφασίζουμε ε, εκ των προτέρων για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί το φάσμα αυτό. Η πολιτική αυτή είναι κάτι που θα εξετάσουμε όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Και κάτι τελευταίο για το φάσμα. οι δυσκολίες σχετικά με την αδειοδότηση είναι πολύ λιγότερες, δεν είναι τόσο ορατές στην πρότασή μας και εσείς το τονίσατε αυτό. Επίσης όσον αφορά την ε, πρόσβαση στις ε, ραδιοσυχνότητες, στις ε, μικρές κυψέλες, είναι επίσης πάρα πολύ πολύτιμη και εμείς επεξεργαζόμαστε τις νέες δυνατότητες του φάσματος και τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα. Ε, επίσης, καλωσορίζουμε και τις ετροπολογίες που επιθυμούν την διατήρηση ορισμένων στοιχείων της ε, πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα για τις ε, επιχειρήσεις και εδώ να απαντήσω και στην κυρία Νίμπλερ, λέγοντας ότι αν ε, ψάχνουμε ανάπτυξη, δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τις τηλεπικοινωνίες, πρέπει να κοιτάμε και τον γενικότερο κλάδο ICT, τεχνολογιών και επικοινωνιών. Και για τον λόγο αυτό η αύξηση της συνδεσιμότητας των επιχειρήσεων είναι κάτι που θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Κάτι τελευταίο επίσης πάνω σε αυτό είναι πως χρειάζεται να εξετάσουμε προσεκτικότερα το πώς οι τροπολογίες ε, αυτές θα ενσωματωθούν καλύτερα στις υπάρχουσες διατάξεις, στο υπάρχον πλαίσιο, έτσι ώστε να επιλέξουμε τα καταλληλότερα μέσα. Τώρα, όσον αφορά το ανοιχτό διαδίκτυο, αυτό είναι κάτι που έχει συζητηθεί διεξοδικά, ιδιαίτερα εν ώψη της ε, επικείμενης ψηφοφορίας στην Επιτροπή ΙΝΚΟ, που είναι και συναρμόδια Αναφέρθηκα ήδη το πρωί σε αυτό και θα πω τώρα σύντομα κάποια πράγματα για ε, το θέμα του σαφούς ορισμού των υπηρεσιών. Αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ως πάρα πολύ σημαντικό και η γλώσσα που έχουμε επιλέξει και η διατύπωση που έχουμε επιλέξει φυσικά δεν πρέπει να είναι ε, μία γλώσσα που καταλαβαίνουν μόνο οι ειδικοί, οι τεχνικοί. Πρέπει να είναι μία γλώσσα που θα καθιστά σαφές ότι πρέπει να υπάρξει σαφής ορισμός των υπηρεσιών, των γενικότερων υπηρεσιών από των διαδικτυακών υπηρεσιών. Και αυτό χρειάζεται να επεξεργαστούν λοιπόν νομικοί, μαθής νομικοί. Κάτι άλλο Τώρα, το αν υπάρχει μια οριστική λίστα των ε, πρακτικών για την διαχείριση της εκκίνησης και αν είμαστε αρκετά ευέλικτοι για να τα εξέλθουμε στις νέες προκλήσεις. Να σας πω ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι φόβοι που έχουν εκφραστεί ότι θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας και η κατάσταση θα γίνει ανεξέλεκτη. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δηλώσει τη στήριξή της στην εισηγήτρια. Θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Τώρα, το θέμα του Μπέρεκ, του Φορέα Ρυθμιστικών Αρχών. Ε, αρχών. Σημεριζόμαστε ότι πρέπει να είναι ισχυρός αυτός ο φορέας και το σύστημα αυτό, το οποίο ήδη έχει αρκετά πλεονεκτήματα, επιδέχεται βελτίωσης. και θα δούμε εάν στο τέλος με την πρότασή μας ο Μπέρεκ αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες. Περιαγωγή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αυτό το εθελοντικό καθεστώς, αυτή την εθελοντική συμμετοχή ήταν κάτι που εμείς θεωρήσαμε πως θα μας έδινε μεγαλύτερη ευελιξία, πως θα δημιουργούσε λιγότερα προβλήματα. Εάν όμως ε, υπάρχει κάτι στο οποίο είμαστε σαφές, σαφείς και ξεκάθαροι, είναι ότι χρειάζεται να συμπεριλάβουμε στην πρότασή μας ότι Πρέπει να αποφύγουμε, να περιπλέξουμε τόσο το σύστημα ώστε να γίνει απρόσιτο για ε, αρκετούς φορείς, για αρκετούς παρόχους. Επίσης ε, και το ζήτημα των εισερχόμενων κλήσεων είναι κάτι που έχει μια απόλυτα λογική εξήγηση, όμως όντως μπορούμε να το αλλάξουμε, μπορούμε να το τροποποιήσουμε. Τέλος, να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Τσίτσεστερ εάν δεν ήμασταν επιμελείς στην απάντησή μας. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Τέλος, όσον αφορά τις ανησυχίες που αφορούν ορισμένες ε, τροπολογίες που διευρύνουν το πεδίο εφαρμογή ε, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έχουμε ήδη αναφέρει σε μια ανακοίνωση το Σεπτέμβριο την άποψή μας σχετικά με αυτό. Δεν χρειάζεται όμως να αλλάξουμε ριζικά τον ορισμό. Και πιστεύουμε πως αυτές οι τροπολογίες είναι τροπολογίες που δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την διεξοδική απάντηση. Για να κλείσει η συζήτηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο, κυρία Καστίγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους. Μεγαλύτερη έκταση, μικρότερη, περισσότερη επικέντρωση, λιγότερη. Όλα αυτά οδηγούν σε μια στάση θετική πιστεύω και επιβεβαιώνει αυτό που είπα και στην αρχή της παρεμβασής μου, ότι δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο, ένα περιθώριο για να καταλήξουμε σε συμφωνία και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας πλήρως και να συνεισφέρουμε έτσι ώστε η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού περάσει από το Κοινοβούλιο, τελικά να καταλήξει σε ένα βήμα πρόοδου προς την ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και της ανάπτυξης της ψηφιακής αγοράς. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα σε καμία παρέμβαση, αλλά θα τελειώσω με αυτό που είπα και στην αρχή, ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας. Και είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να δούμε πέρα από συγκεκριμένα ε, συμφέροντα κάποιων τομέων. Είναι θεμητό όταν γίνονται οι συζητήσεις αυτές, εννοείται πολλές φορές ακούμε και ειδικέ απόψεις που αντιπροσωπεύουν τη μία την άλλη ανησυχία, το ένα ή το άλλο συμφέρον. Ειλικρινά όμως πιστεύω ότι έχοντας παρακολουθήσει τις συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ, την ακρόαση της ε, Ήτρε, της ομάδας μας, φαντάζομαι κι άλλοι έκαναν το ίδιο. Μετά από τη συνεδρίαση που είχαμε για τη μελέτη αντικτύπου που ανέθεσε η Ήτρε για το μακρορυθμιστικό πλαίσιο και την ανάλυση της πρότασης της Επιτροπής, Από όλες αυτές τις συζητήσεις δεν βρήκα άλλο συγκερασμό μεγαλύτερο απόψεων όπως για την ε, κοινωνία των πληροφοριών, για τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την πρόταση. Όλοι όσοι συμμετείχαμε στις συνεδριάσεις αυτές και που ασχολούνται με τον τομέα μπορούν να το επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει τεράστια σύγκληση και προσέγγιση απόψεων για τα περισσότερα θέματα που αναφέρονται εδώ, είτε είναι το ραδιοφάσμα, είτε είναι ο φορέας Μπέρεκ, είτε είναι η περιαγωγή κλπ. κλπ. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, όλοι συμφωνούμε. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι υπάρχει τόσο μεγάλη σύγκληση. Τώρα πιο συγκεκριμένα για κάτι που είπε η Αγγέλικα Νίμπλερ, για κάποια θέματα. Ειλικρινά Αγγέλικα, πώς να πω, πολλά γράφονται, πολλά λέγονται, όχι όμως μόνο για το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε εσύ, αλλά και για άλλα. Και για την κλιματική αλλαγή και για θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιομηχανία, με την ενέργεια, με δικαιώματα και ελευθερίες, ερμηνείες. Για όλα αυτά, κάποιοι τομείς εκφράζονται περισσότερο. Γράφουν σε εφημερίδες, περιοδικά κτλ. Άλλοι εκφράζονται αλλιώς. Πάντως, στη δικιά μας την περίπτωση, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει προσέγγιση, γιατί ξεκινάμε από την ιδέα ότι πρόκειται για ένα παράθυρο ευκαιριών. Ευκαιρίες πρέπει να έχουν όλοι. Το διαδίκτυο δεν είναι τίποτα διαφορετικό από ότι η ζωή εκτός του διαδικτύου, μόνο που εκφράζεται διαφορετικά μέσω μιας τεχνολογίας η οποία επιτρέπει μέσα σε ένα μικροκόσμο, σε ένα οικοσύστημα θα έλεγα, που φτιάχνεται στην κοινωνία με τα χρόνια, δεν αλλάζουμε τις αξίες επειδή χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο ούτε τις οικονομικές μας αξίες. Πιστεύουμε στην οικονομία της αγοράς και μέσα από το διαδίκτυο και έξω από το διαδίκτυο. Θέλουμε τις ευκαιρίες για όλους, τα άτομα, τις επιχειρήσεις και με διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου. Γι' αυτό και οι περισσότεροι από εμά κινητοποιούμεθα, γιατί θέλουμε να προσαρμόσουμε και να διαρθρώσουμε τα πράγματα με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν πρέπει να βάζουμε περιορισμούς. Αντίθετα να είμαστε ανοιχτοί. Έτσι πρέπει να κινηθούμε. Και ειλικρινά πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν δείχνει ένα ανοιχτό πνεύμα και εκφράζει τις αξίες των δημοκρατικών ελεύθερων κοινωνιών και της οικονομίας της αγοράς. Για το ανοιχτό διαδίκτυο, εγώ ακολούθησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πιστεύω ότι είναι μία άποψη καλά ισορροπημένη. Έχουμε τη δυνατότητα να συνονιθούμε λοιπόν μεταξύ μας. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ανοιχτό ίντερνετ, άλλα συστήματα, αλλά είναι θέματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν τώρα ή κάποια στιγμή, αλλά όχι να πάρουμε αποφάσεις που κλείνουν την πόρτα και εμποδίζουν να διευκρινιστούν αυτά τα πράγματα αργότερα ή ανεξάρτητα με το πώς θα διευκρινιστούν αργότερα να έχουμε ήδη προκαταβάλει την κατάσταση παίρνοντας αποφάσεις τώρα. Όχι, πρώτα να διευκρινιστούν αυτά τα πράγματα. Επί της ουσίας αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι σε ένα κείμενο βάζει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς γίνεται. αναγνωρίζει το τι γίνεται στο κείμενο αυτό. Και εμείς δεν λέμε τίποτα άλλο, ούτε προτείνουμε τίποτα που δεν ισχύει σήμερα, που δεν συμβαίνει ήδη. Αυτά. Οπότε, οι δυνατότητες που έχουμε για συμφωνία είναι πολλές. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με το εξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια της γραμματείας της Επιτροπής αυτής. Πραγματικά με στήριξε, με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ειλικρινά δεν έχω λόγια για να το εκφράσω. Έχουν επιδείξει φοβερή επαγγελματικότητα. Ευχαριστώ πολύ και ήθελα να το πω αυτό και δημόσια. E Ακούσαμε λοιπόν όλους ε, σχετικά με αυτή την έκθεση. Η ψηφοφορία, όπως είπαμε και στην αρχή, προβλέπεται για τις 24 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Ευχαριστούμε την Πιλάρα Καστήλιο, τους ε, σκιώδους ηγητές και όλους τους ε, συναντέλφου που συνέβαλαν και θα συμβάλλουν και στο μέλλον στο να ολοκληρωθεί ένα τόσο σημαντικό θέμα. Επόμενο θέμα Πρόκειται για τον υποψήφιο, τον κύριο Νιάση. Αν έχει την καλοσύνη να έρθει εδώ μπροστά, ε, του ευχόμαστε ε, ένα θερμό καλωσόρισμα, το καλωσορίζουμε θερμά. Και όπως ε, γνωρίζετε, ο κύριος Ισβαν Ινιάση προτάθηκε για τον πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική θέση του υποψήφιου διοικητικού διευθυντή του Μπέρεκ. Επιβάλλεται λοιπόν και χαιρόμαστε βέβαια γι' αυτό πριν από τον επίσημο ορισμό του να περάσει και από τη δική μας επιτροπή ε, να κάνει μια δήλωση ο κύριος Σινιάση και κατόπιν να ακολουθήσουν ερωτήσεις και παρεμβάσεις από τους ε, συναδέλφους, οι οποίες και θα απαντήσει. Σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά. Χαίρομαι πολύ για την υποψηφιότητά σας ε, σε αυτή τη θέση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ ε, πόσα πολλά έχετε συμβάλει από τότε που πρωτοπροέκυψε ο οργανισμός αυτός και σας δίνω το λόγο για να ακούσουμε την ομιλία σας, την εισήγησή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη τιμή για μένα που με καλέσατε εδώ για να σας ε, μιλήσω για την υποψηφιότητά μου για το διοικητικό, ε, ως διοικητικό διευθυντή του ΜΠΕΡΕ. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να χωρίσω την εισηγήσή μου σε δύο μέρη. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω, αν κάποιοι ε, θέλουν να βγουν, να βγουν έξω, οι άλλοι να κάτσουν εδώ, έτσι ώστε να μπορεί ο καλεσμένος μας ε, να κάνει την εισήγησή του έτσι εν πλήρη ηρεμία. Παρακαλώ, και όσοι βγείτε, παρακαλώ γρήγορα να βγείτε έξω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα να συστηθώ και μετά να σας ε, αναφέρω γιατί έθεσα υποψηφιότητα για αυτή τη θέση και γιατί πιστεύω πως είμαι ο καταλλήλος υποψήφιος για αυτή τη θέση. Καταρχάς, σε λίγα λόγια για το βιογραφικό μου, για την επαγγελματική μου εμπειρία και για τις σπουδές μου. Είμαι Ούγκρος, όπως ήδη αναφέρθηκε. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην ε, Ανατολική, Βόρειο-Ανατολική Ουγγαρία, κοντά στον ποταμό Τίσα. Τα τελευταία πέντε χρόνια ζω με την οικογένειά μου στις Βρυξέλλες. Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Η κόρη μου βρίσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, ενδιαφέρεται για τις τέχνες, για την ηθοποιία, για τη ζωγραφική. Ο γιος μας ήδη είναι φοιτητή και σπουδάζει πληροφορική, εφαρμοσμένα μαθηματικά, τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν σχέση και με τη μηχανική και έχουμε επίσης και τρεις σκύλους αυτή τη στιγμή στο σπίτι. Προσωπικά είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εκπαιδευτικός. Μετά από κάποια χρόνια εργασίας στον ε, τομέα του management ήθελα να συμπληρώσω τις γνώσεις μου με ορισμένες πρακτικές γνώσεις. Επέστρεψα λοιπόν στα Θρανία, στο ε, Πανεπιστήμιο και έκανα το μεταπτυχιακό μου στη δίκηση επιχειρήσεων. Όταν έγινα δημόσιος υπάλληλος έγινα αφού είχα σπουδάσει στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και πέραν από τα διπλωματικά μου ε, καθήκοντα είχα επιτύχει και στις ε, διπλωματικές εξετάσεις. Η καριέρα μου στις ε, τηλεπικοινωνίες άρχισε το 1990, στις αρχές του 1990, την εποχή των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθερώσης της αγοράς. Και τότε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς άνοιξε η αγορά, η οποία μέχρι τότε ήταν στα χέρια του κράτους. Ήταν επίσης και πολύ ενδιαφέρον ε, το πώς μπήκαν στην αγορά νέοι φορείς. Και εγώ ήμουν ένας από αυτούς, έχει να ε, διευθυντή σε έναν ε, τοπικό πάροχο τηλεπικοινωνιών, ο οποίος μετά από λίγα χρόνια εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του κρατικού παρόχου τηλεπικοινωνιών. 12 λοιπόν χρόνια εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα, περίπου 10 χρόνια σε διοικητικές θέσεις και πιστεύω πως ε, έχω αρκετές γνώσεις του τομέα, του πώς ε, κινείται, του πώς σκέφτονται οι επενδυτές, του τι χρειάζονται οι πολίτες και οι καταναλωτές από τον ε, τομέα των ε, τεχνολογιών και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, εργάστηκα και για κοινοφελείς σκοπούς και πιστεύω πως είναι δυνατόν στον ιδιωτικό ε, τομέα να γίνει αυτό. Έπειτα τον μεταπίδησα στο δημόσιο, στο αρμόδιο Υπουργείο, Υπουργείο Τεχνολογίων Τηλεπικοινωνιών. Απέκτησα, πιστεύω, μια πολύ καλύτερη κατανόηση όχι μόνο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όσοι χαράσουν την ε, πολιτική τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών, αλλά και το πώς ε, λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Και πιστεύω πως ε, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, στα κατημέλη σε, αυτή, σε αυτό το χώρο. Έπειτα, όταν η Ουγγαρία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργάστηκα εκεί, εργάστηκα στην Προεδρία και ήταν εξαιρετική εμπειρία, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία που προσέθεσε πιστεύω στις γνώσεις μου και ήταν επίσης και τιμή μου που εργάστηκα στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και προείδρευσα σε αυτές. Μέσω της εργασίας μου αυτής ε, απέκτησα βαθιές γνώσεις του πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς ε, εκτιλήσεται η νομοθετική διαδικασία. Από το 2005 λοιπόν, από την ένταξη της, ε, λίγο μετά την ένταξη του Ουγγαρίας και μετά, απέκτησα ε, βάθος γνώσει πολλών ε, τομέων ε, σχετικών με τις ε, τεχνολογίες, για παράδειγμα της νομοθεσίας σχετικής με την περιαγωγή. Θεωρώ μεγάλη πρόκληση την θέση αυτή του διοικητικού διευθυντή του Μπέρεκ. Πιστεύω πως η επαγγελματική μου εμπειρία, οι σπουδέ μου και οι μέχρι τώρα γνώσεις μου και η προσωπικότητά μου θα αποτελέσουν προσόν για τον Μπέρεκ και για την θέση αυτή θεωρώ πως η θέση αυτή μου ταιριάζει. Μου ταιριάζει όχι μόνο λόγω του πρώτερου επαγγελματικού βίου μου, αλλά πιστεύω πως μπορώ να συνεισφέρω σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρω πως η θέση αυτή είναι πάρα πολύ υπεύθυνη και πρέπει να συνδυάσει και διοικητικά ε, και διπλωματικά καθήκοντα, αλλά και management και έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, διότι διαχειρίζεται πόρους, κονδύλια και ταυτόχρονα πρέπει να συνδυάσει και, το, και την παροχή των υπηρεσιών. Ο κύριος στόχος φυσικά είναι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου και αυτή είναι και η κύρια αποστολή του Μπέρεκ εξάλλου. Και στον κανονισμό λειτουργίας του Μπέρεκ αναφέρονται με σαφήνεια οι προτεραιότητες και οι αρμοδιότητες και πιστεύω πως ε, θα συνεισφέρω στην καλύτερη εφαρμογή των στόχων και του, της αποστολής του Μπέρεκ. διότι ο Μπέρεκ εργάζεται για κάτι το οποίο εσείς θα κληθείτε μετά να εγκρίνετε, να ψηφίσετε. Ε, το πακέτο που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή είναι το πακέτο των τηλεπικοινωνιών για την ενιαία αγορά και εσείς έχετε ένα και σημαντικότερο ρόλο και ελπίζουμε στην στήριξή σας στο Νμπέρε και στο έργο του. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι με την ιδιότητά μου, αυτή ως ε, διοικητικός διευθυντής, εάν ε, εκλεγώ, θα εργαστώ στην αναδιοργάνωση του γραφείου και στην βελτίωση της αποδοτικότητάς του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτά από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμεί σα ευχαριστούμε για την, ε, την παρουσίαση των προσόντων σα. Και τώρα λοιπόν ε, ξεκινούν οι παρεμβάσεις. Πάλι κυρία Καστήλιο, εκ μέρου ε, του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να απευθυνθώ στον, πώς να το πω, υποψήφιο διοικητικό διευθυντή του Μπέρεκ. Καλώς ήρθατε. Χτες είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε οι δυο μας. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί η θέση σας. Όπως γνωρίζουμε, έχει μακρά εμπειρία στα θέματα αυτά. Και φτάνει σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή. Υπάρχουν τα θέματα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπάρχει το BEREC και κυρίως γι' αυτό το τελευταίο η Επιτροπή μας έχει οθετήσει θέση σαφώς υπέρ της διατήρησης και της παγίωσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φορέων Ρυθμιστικών Αρχών. οργανισμός, στην σύντομη ζωή του μέχρι σήμερα κάνει σημαντικό έργο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το ΠΕΡΕΚ έχει έναν ρόλο τον οποίο φέρνει πολύ καλά σε πέρας αλλά πολύ πιθανόν να χρειαστεί να αναλάβει και άλλο ρόλο, συντονιστικό για παράδειγμα, για άλλε σημαντικέ πτυχές που έχουν να κάνουν με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την κοινωνία των πληροφοριών, τι τεχνολογίε πληροφοριών δηλαδή. Έχει ένα προφίλ που προσαρμόζεται πολύ καλά στην εμπειρία και στις αρμοδιότητες. Νομίζω ότι ο κύριος Ισβανινιέσκη και από το βιογραφικό του και από την εμπειρία του φαίνεται ότι είναι κατάλληλος για να αναλάβει τη θέση αυτή του διοικητικού διευθυντή του Μπέρεκ. Ελπίζουμε όντως να πετύχετε. Σε πολλούς τομείς έχει να παίξει σημαντικό ρόλο ο Μπέρεκ και αυτό το είπανε πολύ εδώ. Φάνηκε αυτό. Τίποτα άλλο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε, συνάδελφο Χέρτσοκ. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Φαίνεται ότι σήμερα είναι η μέρα μου. <laughs> Μιλάω για τρίτη φορά. Στην Ήτρε, βέβαια. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά ε, πολύ καλά έκανα και έμεινε εδώ και συμμετέχω και στη συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω για τον κύριο Ιγνέτσι με πολύ λίγα λόγια και κατόπιν να μιλήσω για τον ίδιο τον οργανισμό τον Μπέρεκ. Γνωρίζω τον Λάσλο όσο είμαι μέλος του Κοινοβουλίου. Ήρθαμε σχεδόν μαζί εδώ και νομίζω ότι το γεγονός ότι σε μία διαιρεμένη χώρα όπως είναι η Ουγγαρία ο Λάσλο χέρι της υποστήριξης όλων, από όλε τι πλευρές και αυτό μιλάει από μόνο του. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα επί των οποίων θα μπορούσαν να συμφωνήσουν τα βασικά κόμματα της Ουγγαρίας, το Σοσιαλιστικό και το Χριστιανοδημοκρατικό, αλλά εδώ συμφωνούν όλοι σχετικά με την ε, προσήλωσή του που μέχρι τώρα ωφέλησε και τη χώρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια ε, όσο συζητιόταν το πακέτο τηλεπικοινωνιών μετά την Ουγγρική Προεδρία και αργότερα και με τα γενέστερα ο Λάσλο αποδείχτηκε κάποιος που είχε απάντηση για όλα. Και νομίζω αυτό το είπαν όλες οι εταιρείε που συνεργάστηκαν με την Ουγγρική Προεδρία. Επίσης, είναι ενδεικτικό ε, το ότι εδώ έχουμε και την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου, το οποίο είναι γνωστό για το ότι είναι σκληρό στις ακοράσεις του. Και επιτρέψτε μου για λίγο να μιλήσω για τον οργανισμό Μπέρεκ. Μιλήσαμε για τον οργανισμό αυτό και προηγουμένως και είναι σαφές ότι φορείς όπως είναι ο Μπέρεκ σαφώς και χρήζουν πολλών βελτιώσεων. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, ήμουν σκιώδης ηγήτρια για τους οργανισμούς ε, επανειλημμένα συνέβη αυτό και θέλω να πω απευθυνόμενοι καταρχήν προς τους ε, συναδέλφους ότι όλοι οι οργανισμοί τα πρώτα πέντε χρόνια έχουν αντιμετωπίσει μία πρόκληση διότι ε, τους ανέθεσε κάποια θέματα το Κοινοβούλιο, αλλά όχι με απόλυτη σαφήνεια. Το Συμβούλιο έχει επιλέξει την έδρα τους και εκεί πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα, μερικές φορές υπάρχουν τα γραφεία, δεν υπάρχει το προσωπικό ή υπάρχει το προσωπικό και δεν υπάρχουν ε, τα γραφεία. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Έτσι λοιπόν από την ύπαρξη των οργανισμών αποδεικνύεται ότι από τους 60 περίπου παρεμφερείς οργανισμούς που έχουμε ε, όλοι αυτοί οι οργανισμοί τα πρώτα πέντε χρόνια περνάνε από τις παιδικές ασθένειες και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό ε, γιατί δεν πρέπει να αλλάζουμε και συνεχώς να ξαναλάζουμε τις αρμόδιότητες αυτών των οργανισμών ε, τα πρώτα πέντε χρόνια. Κυρίως να μην το κάνουμε κατά κόρον, ε, διότι λέμε ότι ακόμα δεν λειτουργούν αποτελεσματικά ή διότι υπάρχει κάτι που χρήζει βελτίωσης. Και επιτρέψτε μου και μία ερώτηση προς τον κύριο Ιγνάση σχετικά με το πώς ακριβώς επιθυμεί να συνεργαστεί με άλλους ε, παρεμφερείς οργανισμούς, με εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές, ε, έτσι ώστε να μην χάνουμε χρόνο με περιττές αναδιοργανώσεις, ανταυτού να αναζητήσουμε τη βελτίωση. Και η βελτίωση, κατά την άποψή μου, μπορεί να είναι προς την εξής κατεύθυνση ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν καλύτερες υπηρεσίες καλύτερη ψηφιακή πρόσβαση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τον οργανισμό Μπέρεκ και νομίζω το Κοινοβούλιο είναι ανοιχτό σίγουρα. Κύριε Γνάτση, δεν, ελπίζω να μην είναι αυτή η τελευταία σας επίσκεψη εδώ, ε, να είναι η πρώτη ε, με το καινούργιο αξίωμά σας και ελπίζουμε να επανέλθετε. Οποτεδήποτε έχετε να μας πείτε κάτι, εμείς θα έχουμε ανοιχτά αυτιά. Σας ευχόμαι καλή τύχη και χαίρομαι που έχουμε κάποιον που γνωρίζει την αγορά τους κύριους παρόχους, ε, έχει ανοιχτό μυαλό, μια πολύ καλή προσέγγιση, κάποιος ε, που είναι σε πολύ καλή θέση διοικητική και νομίζω είστε πραγματικά η τέλεια επιλογή για τη θέση που συζητάμε. Είτε... Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος. Ε, το λόγο να λέω τον Ντενόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι Με μεγάλη μου ευχαρίστηση βλέπω ότι ο κύριος Συχνές είναι ο κύριος υποψήφιος για αυτή τη θέση και καταλληλότερος, διότι πιστεύω ότι η εμπειρία του ε, είναι η κατάλληλη και θα μπορέσει να συνεισφέρει στην καλή λειτουργία του Μπέρεκ. Μπορούν να μας φαίνονται πολύ εύκολα αυτά που γίνονται εκεί. Στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ δύσκολο να μπορεί κανείς να συνδέει όλα αυτά, το νομοθετικό έργο να έρχεται σε επαφή με ε, τους ε, ρυθμιστικούς φορείς. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχηθώ στον ε, κύριο Ιγνέση καλή αρχή, καλή επιτυχία στο έργο του. Ο τομέας των ε, τηλεπικοινωνιών είναι ένας ταχύτατα εξελισσόμενος τομέας έχει μεγάλη δυναμική και είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρούμε τις ε, εξελίξεις, τις πολύ γρήγορες εξελίξεις, ε, οι οποίες είναι τόσο γρήγορες που δεν τις προφταίνει πολλές φορές η νομοθεσία. Και αυτό επειδή τα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται είναι περίπλοκα. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να ακολουθεί η νομοθεσία την ταχύτητα των εξελίξεων. Μία πολύ απλή ερώτηση έχω. Εσείς πώς φαντάζεστε την συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ο τομέας αυτός, όπως ε, είπα και πριν, έχει ταχύτατες εξελίξεις, μεταβάλλεται συνεχώς και η συνεργασία λοιπόν με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν θα είναι εύκολη. Και κάτι άλλο εύχομαι να ασκήσετε τα καθήκοντά σας με επιτυχία. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς και χαίρομαι πάρα πολύ που κάποιος με τα δικά σας προσόντα λαμβάνει μια τέτοια θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άντερς Ντότερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Ιγνάτσα στην Επιτροπή Βιομηχανίας και να τον συγχαρώ για την υποψηφιότητά του για τη θέση του διοικητικού διευθυντή του Μπέρεκ. Υπάρχουν εκκρεμότητες στον, στην νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες. Ιδιαίτερα η οδηγία 2258 είναι μια οδηγία η οποία διχάζει τα κράτη-μέλη. Και από ό,τι έχω δει μετά από τον καιρό που βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο, η συνεργασία ανάμεσα στις αρχές προστασίας δεδομένων και τα κράτη-μέλη είναι αρκετά καλή. Έχουμε λιγότερη ανάγκη για συντονισμό μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και περισσότερη ανάγκη για διάλογο ανάμεσα στον ΠΕΡΑ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διάφορες αρμοδιότητες ε, που έχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εσείς πώς θα διευκολύνετε το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών ε, αρχών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και επαρκής εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσατε ίσως να μας αναφέρετε κάποιες από τις περιπτώσεις πλοκές, κάποιες από τις δυσκολίες που θα προκαλέσει ο νέος αυτός κανονισμός. Τουλάχιστον στη Σουηδία, στη χώρα μου, θα ε, προκαλέσει μια σύγχυση σχετικά με το ποιος θα, ποια αρχή είναι αρμόδια όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, άλλες ερωτήσεις. Όχι. Μπορείτε τότε, κύριε πάρετε το λόγο και να απαντήσετε σε ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σας και για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Με χαρά μου βλέπω ότι εκτιμάτε το έργο και τα επιτεύγματα του Μπέρεκ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα σχόλιά σας, αλλά και από τις συζητήσεις που είχαμε για το πακέτο τηλεπικοινωνιών μέχρι τώρα και από την περισσυνή αξιολόγηση του Μπέρεκ και του έργου του Μπέρεκ. Έχω λοιπόν ε, λάβει καλά μηνύματα από αυτό και θα το μεταφέρω και στους υπόλοιπους ε, συναδέλφους το, του Μπέρεκ. Τώρα όσον αφορά τις ερωτήσεις που μου θέσατε, ε, κύριε Τοσενόφσκι και κυρία Άντερς Ντότερ, με ρωτήσατε παρόμοια περίπου πράγματα σχετικά με την ε, συνεργασία και πώς θα εγώ θα διευκολύνω τη συνεργασία ε, των ε, ρυθμιστικών αρχών. Σωστά είπατε ότι ο ΠΕΡΕΚ είναι μια πολύ ειδική υπηρεσία, είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία και κύριο έργο του, κύριε αποστολή του ΠΕΡΕΚ, είναι η διευκόλυνση της ε, συνεργασίας αυτών των ομάδων επιρρογνωμόνων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και συνεργασία στους διάφορους τομείς και η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Αυτή είναι η κύρια αποστολή του Φορέα Ρυθμιστικών Αρχών. Και η οδηγία 2258 που ανέφερε η κυρία Άντερ Στότερ υπάγεται στις αρμοδιότητες του Μπέρεκ. Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι δεσμεύομαι για το ότι ο Μπέρεκ θα συνεχίσει να προσπαθεί για την καλή συνεργασία και την βελτίωση των ήδη ε, υφιστάμενων δομών. Μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο το τι κάνουμε, πώς ε, τα κάνουμε, τι εξελίξεις υπάρχουν και πώς προχωρά το κάθε θέμα, η κάθε οδηγία, ο κάθε φάκελος. Κυρία Χέρτσογκ, με ρωτήσατε πώς θα βελτιωθεί η συνεργασία και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ οργανισμών. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο Μπέρεκ πιστεύει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αυτό κάνει. Και είναι καλό αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το, την ιδιότητα αυτή της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και να αντλήσουμε από αυτές έτσι ώστε να οργανώσουμε τη λειτουργία μας ακόμα καλύτερα. Να πάρουμε λοιπόν θετικά στοιχεία από άλλους οργανισμούς που έχουν ήδη περισσότερη εμπειρία και θα μπορούσαν να μας συμβουλεύσουν και να μας ε, στηρίξουν στις προσπάθειες για βελτίωση αυτές. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να έρθω εδώ, να σας ευχαριστήσω και για τη μεγάλη στήριξη που έλαβα από εσάς και για το πρόσωπό μου και για το Μπέρεκ. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι στο μέλλον θα είμαι πάντα διαθέσιμος για εσάς. Σας συγχαίρω και εγώ και εγώ συμφωνώ με τα συγχαρτήρια. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη και ελπίζουμε τελικά όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ικανοποιητικά. Καλή δουλειά σας εύχομαι και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Δεν νομίζω ότι θα χαθούμε. Abbiamo ancora un punto da affrontare, che sarà molto breve peraltro. Λοιπόν, πάμε λοιπόν ε, στο θέμα του backloading, το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένα και τα μέλη της Επιτροπής μας, ε, όπως προβλέπεται η διαδικασία, εκλήθησαν να ορίσουν μια συγκεκριμένη μερομηνία, συγκεκριμένα στις 24 Ιανουαρίου για να καταθέσουν μέχρι τότε τις αντιρρήσεις τους. Και έχουμε λοιπόν ε, διατύπωση αντιρρήσεων από τακτικά μέλη και αναπληρωτές ε, έτσι λοιπόν ε, θα υπάρξει η ψηφορία αύριο. Σήμερα θα συζητήσουμε ε, προκατακτικά για την ε, αυριανή ψηφοφορία. Η συζήτηση θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ένα, το πολύ δύο λεπτά αναπολιτική ομάδα Πρώτα η συνάδελφο Τζόρνταν θα μας ε, παρουσιάσει τις αντιρρήσεις ε, και αν θέλουν ε, οι άλλες πολιτικές ομάδες μπορούν και αυτές να τοποθετηθούν και έτσι θα κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα θα παραπεμφθεί για αύριο. Εκεί θα ψηφίσουμε. Η κυρία Τζόρνταν έχει το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα εννέα ευρωβουλευτές που έχουν υπογράψει την πρόταση και μου ζήτησαν να παρουσιάσω την ε, θέση τους, οπότε θα σας διαβάσω αυτό που μου είπαν. Το, τα μέτρα της μείωσης του όγκου για το 2014 μέχρι το 2016 δεν είναι αναγκαία έτσι ώστε να επιτύχουμε το στόχο της οδηγίας, στόχος ο οποίος έχει να κάνει με την μείωση των ε, προκαθορισμένων ορίων εκπομπής του θερμοκηπίου η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στον ε, καλό δρόμο για την μείωση των εκπομπών αερίων μέχρι το 2020. Το κύριο μέσο που σχεδιάστηκε, σχεδιάστηκε έτσι ώστε η ίδια η αγορά να αυτορυθμίζεται για, τον, ε, για την επίτευξη του στόχου της μείωσης χωρίς παρεμβάσεις από αρχές και χωρίς τεχνητές ε, αλλαγές στην, στην τιμή των επιστοποιητικών. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο ναι, να επιτύχουμε την όσο το δυνατόν ομαλότερη λειτουργία του συστήματος ETS. Ε όπω σα είπα, εγώ δεν το υπέγραψα, δεν υπέγραψα την αίτηση αυτή, όμω τη στηρίζω απόλυτα. Έτσι λοιπόν αύριο θα έχετε μία ακόμα τουλάχιστον υπογραφή τη δική μου. Και θα ήθελα να πω ότι κοίταξα έτσι πολύ γρήγορα την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που έφτασε σήμερα για την ενεργειακή πολιτική από το 2020 και μετά και βασισμένη στην πρόταση αυτή είμαι ακόμα πιο σίγουρη για τις αντιρρήσεις μας σχετικά με το backloading. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τα ίδια λάθη με την πρόταση του 2020, τώρα στην πρόταση για το 2030. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, δεν μιλήσατε, δεν υπογράψετε βέβαια, αλλά από ό,τι κατάλαβα... Ε, υπερασπιστήκατε σωστά αυτή την ένσταση. Τάρια, del ALDE. ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στο τι ακριβώ κάνουν αυτές οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Πιστεύω πως αυτή δεν είναι η στιγμή για όποιους ε, δεν θεωρούσαν καλό όλο το σχέδιο του backloading να το σταματήσουν. Διότι η συζήτηση για το backloading έχει γίνει. Έχει γίνει επίσης και η πρώτη πρόταση. Η δεύτερη πρόταση, την οποία ενέκριναν 27 κρατημέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία, την δεύτερη φορά. Και δεν νομίζω πως Παρότι σέβομαι τις απόψει των ε, συναδέλφων, δεν νομίζω πως ε, πρέπει να σταματήσουμε αυτές τι πράξει εξουσιοδότησης μόνο και μόνο επειδή εσεί διαφωνείτε. Ο μόνος εδόκιμος λόγος ε, είναι επειδή δεν σας αρέσει η πρόταση της Επιτροπής για το 2030. Έτσι λέτε εσείς. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ο μόνος δόκιμος λόγος είναι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπερνά τις αρμοδιότητές της, ξεπερνά τις εξουσίες της με την πρόταση αυτή. Και σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο εδώ. Είναι ένα ξεκάθαρο πολιτικό ε, μήνυμα από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι το Συμβούλιο θέτει τις ε, προϋποθέσεις, τα μέτρα για, ε, που απαιτεί αυτή η πολιτική απόφαση. Και καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν εδώ να, να τοποθετηθούν πολιτικά και να δώσουν το στίγμα τους και δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουν. Όμως εμείς δεν μπορούμε να ε, φέρουμε αντίρρησης για αυτή την πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους λοιπόν τώρα των Σοσιαλδημοκρατών. Κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η συζήτηση για το backloading είναι κάτι που ψηφίσαμε, στηρίξαμε. Δεν νομίζω ότι τώρα πρέπει να ανοίξει και πάλι η συζήτηση. Είναι σαν να προσπαθούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση από την πίσω πόρτα. Η ομάδα μου θα είναι κατά της απόρριψης των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Θα ψηφίσουμε όχι στο ψήφισμα. Για να είμαστε συνεπείς. Νομίζω ότι είναι σαφής η θέση των σοσιαλιστών από αυτού. Ο συνάδελφος Τσίτσεστερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Και εμείς θα είμαστε συνεπείς με την πρώτερη θέση μας. Εγώ υπέγραψα την πρόταση αυτή. Τη στήριξα στηρίζω και την επιχειρηματολογία που ακούσαμε από την κυρία Τζόρνταν. Και θα προσθέσω μάλιστα ότι πιστεύουμε ότι είναι ένα δυσανάλογο μέτρο το οποίο δεν είναι αναγκαίο. Είναι άλλη μια περίπτωση που προσπαθεί η Επιτροπή να βρει μια λύση σε ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει. Και δεν χρειάζεται. Το λένε στο κάτω-κάτω εφόσον μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας για το 2020. Είναι θέμα αναλογικότητας. Βέβαια, εγώ δεν βλέπω γιατί να μην ξανανοίξει το επιχείρημα. Είμαστε σε μια δημοκρατία και κανείς έχει το δικαίωμα να διαφωνήσει με την πλειοψηφία. Ελπίζω, έτσι. Ακόμα και αν υπάρχει μια πλειοψηφία, έτσι, κύριε Μαντουρέλ. Τι λέτε, ότι είσαστε υπέρ της λογοκρισίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε, κύριε Τσίτσεστερ. Πάντα πνευματόδης η συνάδελφος Ιμπνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από την αρχή έχω την αίσθηση ότι η ανάμιξη στο σύστημα ποσοστώσεων εκπομπών ερήνων του θερμοκήπη είναι κάτι που μας κάνει να διαπιστώσουμε ότι μην αλλάζοντας τα πράγματα δεν βελτιώνεται η κατάσταση ούτε για τη βιομηχανία ούτε και για κανέναν άλλον. Η επικέντρωση είναι κακό για τη βιομηχανία και πρέπει να δούμε λιγάκι τι γίνεται και με τη βιομηχανία εκτός Ευρώπης. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις βιομηχανικές οι οποίες φεύγουν από την Ευρώπη. πάνε στη Λευκορωσία ας πούμε. Συνεπώς, το πάγωμα των ποσοστώσεων με πλειοψηφία, εντάξει μπορεί να υπάρχουν αρκετοί από εμά που το θέλουν, αλλά τελικά τι θέλουμε στην πραγματικότητα, θέλουμε να καταστρέψουμε το σύστημα. Ή θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις ποσοστώσεις, μα δεν πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν λειτουργεί το σύστημα να μην κάνουμε μόνο μικρές αλλαγές, αλλά να κάνουμε σε βάθος μεταρρύθμιση. Συμφωνώ ότι δεν φτάνει. Όσο για τις ή πράξεις, δεν βοηθούν εδώ. Αντίθετα, δημιουργούν και κάνουν ζημιά στις βιομηχανίες μας. Ευχαριστούμε. Πάντα είναι καλό να έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε, έτσι. Εκπρόσωπο της Επιτροπής θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα παρακαλώ, έτσι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, θα είμαι σύντομη γιατί έχουν γίνει ήδη πολλές συζητήσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Όπως είπαν και άλλοι, οι εκτελεστικές εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν πει ότι εντατικά χρησιμοποιείται το backloading, ότι το παρακολουθούμε αυτό και στην Ευρωπαϊκή τον Επιτροπή τον τελευταίο μήνα. Είπαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να υποβάλουν έσταση εφόσον διαπιστώσουν ότι ξεπερνούνται οι εξουσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις καταξιδότητε πράξεις. Το σύστημα αυτό εμπορίας ε, εκπομπών είναι πετυχημένο. Στόχος τη οδηγία στο παράρτημα 1 είναι σαφής. Λέει αποτελεσματικές μειώσεις εκπομπών και λαμβάνοντα υπόψη και το μακροπρόθεσμο το μέλλον, δηλαδή μετά το 2020. Δεν υπάρχουν νομικέ βάσεις για να αντιταθούμε στην πράξη αυτή και επί τη ουσία πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο το backloading, δηλαδή ο πιστοβαρή προγραμματισμός, γιατί χρειάζεται μερικέ φορές επειδή είναι πολύ χαμηλέ οι τιμέ και τότε υπάρχει ο κίνδυνος να δοθεί το μήνυμα το στραβό από τις τιμές, ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και ότι θα συνεχίσουν οι εκπομπές μακροπρόθεσμα, συνεπώς η βιομηχανία μπορεί να πάρει αποφάσεις οι οποίες τελικά να επιβαρύνουν περισσότερο τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Καλώς πήρανε όλοι το λόγο σε θέλω να θα ψηφίσουμε αύριο για αυτό το θέμα. Έτσι ολοκληρώνονται οι εργασίες της Επιτροπής μας. Στις 5.30 θα αρχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών και η συνάδελφος τότε θα προεδρεύσει. Εντάξει, αύριο θα ξαναβρεθούμε για τις προφορίες.